νέο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις της κυρίας Μάλστρομ εξ του Συμβουλίου. Mrs. Minister, you Έχετε το λόγο κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, άργησα λίγο να, ακούσω την ε, μετάφραση των λέγατε. Κυρία Άστον, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το πρόβλημα που τώρα αντιμετωπίζουμε ε, προκειμένου είναι το ίδιο όπως και στον υπόλοιπο κόσμο ε, εξτρεμισμός και τα ναρκωτικά τα οποία από το Αφγανιστάν εύκολα καταλήγουν στους δρόμους της Ευρώπης, στις πιάτσες όπου και γίνεται η ανάγκη να δούμε πώς δεν θα είναι ασφαλή καταφύγια για το οργανωμένο έγκλημα αυτές οι δύο χώρες, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Έχει ελκύσει την ε, προσοχή το Αφγανιστάν βέβαια, διότι πάρα πολλές χώρες εκεί έχουν εμπλακεί, έχουν δεσμευτεί, έχουν στείλει στρατό, αλλά και στο Πακιστάν οι προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές και η επίλυση του προβλήματος του Αφγανιστάν εξαρτάται από το τι πορεία θα πάρουν τα πράγματα στο Πακιστάν. Δηλαδή είναι αυτές οι χώρες αλεξαρτώμενες σε πολλά. Μας ζήτησαν να κατεβάσουμε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και για αυτό και εμείς συντάξαμε αυτό το πρόγραμμα δράσης σαν κείμενο το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογο αυτό σαν μέσο πολιτικής. Επομένως, θα πρέπει και στη συνέχεια να προσαρμόσουμε ό,τι ίσχυε προηγουμένως και να αναπροσαρμόσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Έχουμε στα πλαίσια αυτά επισημάνει κάποιες προτεραιότητες να δούμε πώς θα είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Ε, επομένως, εδώ επισημαίνεται τι θέματα πρέπει να προσέξουμε, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα επίση στου ανθρώπου τη περιοχή, ότι θα είμαστε συνεπεί προς όσοι έχουν προσχεθεί. Ε, Για αυτό σα λέω ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες και ότι μια απο τι κορυφαίε προτεραιοτητες και οτι μια που το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μια κρίση με καμπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι γίνανε οι εκλογέ, χωρί να είναι βέβαια ιδανική η κατάσταση που εκεί επικράτησε κατά τι εκλογέ. Επίσης, προτιθέμεθα να στηρίξουμε τους Αφγανούς για την πορεία που έχουν κάνουν, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση που συγκροτήθηκε, να τη βοηθήσουμε στο πρόγραμμα που κατήρθησαν, να τους φέρουν πιο κοντά στη διεθνή κοινότητα. Ο πρόεδρος Καρζάη, επί την των καθηκόντων του, έκανε κάποια ομιλία που έδωσε κάποια θετικά μηνύματα και είπε ότι προτίθεται να ανανεώσει τους δεσμούς του με τον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε εμείς θέλουμε να υπάρχει ε, δυναμική διακυβέρνηση γιατί δεν θέλουμε άλλη μια πενταετία να πάει χαμένη χωρίς να υπάρξουν κάποια θετικά βήματα πρόοδου. Θα πρέπει επομένω το κράτος εκεί να συγκροτηθεί, να δεσμευθεί όσον από τη διεθνή κοινότητα, Και επίσης σας επισημαίνω ότι οι Αμερικανοί του χρόνου θα στείλουν 30.000 30.000 προσωπικό για να προσταθούν σε αυτούς που ήδη υπάρχουν στη χώρα και το ίδιο θα κάνουν και άλλοι σύμμαχοι τουλάχιστον άλλοι 7.000 θα σταλούν πέραν των υπαρχόντων εκεί προσώπων που ανέρχονται στις 30.000 και μιλώ για στρατιωτικούς και πολιτικό προσωπικό Άρα, αν δεν υπάρξει εκεί ένα πλαίσιο σταθερότητας και χρηστής διακυβέρνησης, δεν είναι δυνατόν να απόσυρθούν τα στατεύματα από τη χώρα αυτή. Δηλαδή να πρετανεύσει το κράτος δικαίου, να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Δεν είναι επομένως μόνο θέματα ασφάλειας. Σωστή διακυβέρνηση χρειάζεται να ξεκινήσει κάποιος ρυθμός ανάπτυξης έχουμε δεσμευτεί όσον αφορά αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει όμως και οι ίδιοι οι Αφγανοί να καταλάβουν ότι πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, γιατί είναι δική του κυβέρνηση και αυτοί έχουν λάβει την βελτίωση της κατάστασης της χώρας. Οπότε θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αρχίσει να υπάρχει εμπιστοσύνη προ του ηγέτε τη χώρα. Αυτή η αφγανοποίηση να αρχίσει να συνεχιστεί και η Ένωση βέβαια να βοηθήσει όλο ένα και περισσότερο την κατάσταση. Να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα της χώρας. Σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο. Χρηστή διακυβέρνηση, καταπολέμηση της διαφθοράς, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βέβαια είναι σημαντική για ανάπτυξη της γεωργίας. Να εξασφαλιστεί ο, το ότι όλοι αυτοί οι Αφγανοί που είναι πλειοψηφία και μένουν στην Ήπεθρο θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Να δούμε επίσης πώς θα βρούμε κάποιο διέξοδο για τους παλαιούς πολεμιστές τώρα θα πρέπει φυσικά να βρουν κάποιο ελληνικό τρόπο να κερδίσουν το ψωμί τους. Το 2008 ξαναρθεί η δημοκρατία στη χώρα. Αυτός ο δημοκρατικός μετασχηματισμό ήταν εντυπωσιακό, όμω παρόλα αυτά είναι ευάλωτη η κατάσταση. Φυσικά στο, στη χώρα, στο Πακιστάν λέμε, οι Ταλιμπάν αποτελούν έναν κίνδυνο. Είχαμε διάφορες ε, ε, επιθέσεις αυτοκτονικές βομβιστών Άρα να βοηθήσουμε και τη χώρα εκείνη ακολουθώντας τις συστάσεις του Μάικλ Γκάλλαρ του 2008. Είχε τότε φτιαχτεί ένα βασικό πλαίσιο για να βοηθήσει τη χώρα να σταθεί στα πόδια της να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση το Πακιστάν σε συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση να βρει μια συνέχεια η συνάντηση κορυφής του Ιουνίου του 2009 και έτσι βοηθώντας τα νόμιμα θεσμικά όργανα θα προχωρήσει η δημοκρατία, θα καταπολεμηθεί ε, το λαθρεμπόριο, το εμπόριο των εργοτικών και έτσι το κράτος να σταθεί στα πόδια του και να αρχίσει να λειτουργεί εύρεθμα. Οι ίδιοι οι Πακιστανοί να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στη χώρα τους ασφάλεια και σταθερότητα και να καταπολεμηθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας. Ακόμα και εκείνοι που έχουν το στατοπεδό τους στο Πακιστάν και επιχειρούν στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τις δεσμεύσεις μας. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει η χώρα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και το ίδιο ισχύει και για τις δύο χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις σημαντικές σε αυτές τις δύο χώρες. Ήδη έχουν επιτευχθεί πολλά και στις δύο αυτές χώρες. Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν πέτυχαν πολλά από μόνα τους, από μόνες τους αυτές οι χώρες, αλλά και η διεθνή κοινότητα επίσης. Έχουμε χαράξει κάποιες στρατηγικές, αλλά τώρα με κάποια πρακτικά επιτόπου μέτρα θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία σχεδιάσαμε. Το λόγο θα πάρει η κυρία Άστον εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mrs. Um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώ με το Αφγανιστάν. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή των σχέσεων μας. Θα πρέπει η κυβέρνηση να τίνει ευήκονους τις ανάγκες των, του Αφγανού λαού. Και πρέπει να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση αυτή, αλλά και να επηρεάσουμε τα πράγματα. Η διεθνή διάσκεψη, η πρώτη διεθνή διάσκεψη μια σειρά, ξεκινάει ε, τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο. Η Κομισιόν αυξάνει ε, στα 200 εκατομμύρια ευρώ ε, την βοήθειά της πόρους που χρειαζόμαστε για τον τομέα της υγείας, για θεραπευτικές αγωγές προς τις ε, γυναίκες αλλά και τα κορίτσια. Επίσης εκρίζωση της καλλιέργειας παπαρούνας. Αυτά όμως είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στα πλαίσια μιας συντονισμένης διεθνούς απόκρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι Αφγανοί θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ΑΕΕ. Το σχέδιο δράσης του Οκτωβρίου μας δίνει δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Μαζί με τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα στην περιοχή αυτή του κόσμου αλλά και στη εθνική κοινότητα για την αποφασιστικότητά μας. Επίσης, υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες του Πρόεδρου Καζάη ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το σχέδιο δράση επιβεβαιώνει ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου και την γεωργία. Ήδη βοηθάμε στην Καμπούλ προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε τώρα να εξαπλώσουμε τη βοήθειά μας και στις διάφορες επαρχίες της χώρας ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει και εκεί α, το κράτος. Και είναι ευτυχές το γεγονό ότι οι α, διαφωνούντες πλέον έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν. Θα ήθελα να αποτύσω φοροτιμή στον κύριο Μπέρμαν και, την, και το επιτελείο του για, μια, για ένα πολύ καλό έργο υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης και δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθεί αυτό που έγινε με τις εκλογέ. Επίσης, επιτόπου <clears throat> θα έχουμε δράσεις, συνεργασία με τα κράτη-μέλη και ελπίζω να συντονίσουμε τις προσπαθίες μας τόσο ώστε να έχουμε μια συνεκτική και συνεπή αντιμετώπιση. Για το Πακιστάν τώρα. Η βασική μας ανησυχία αλλά και μέρημνα είναι μια σταθερή δημοκρατία χωρίς τρομοκρατία το σχέδιο δράσης το υπογραμμίζει αυτό σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ιουνίου συμπεριλαμβάνει θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης και ενίσχυση για το εμπόριο και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εφαρμογή των συστάσεων ε, της ε, αποστολής ε, παρατηρητών με τις εκλογέ του 2008. Έχουμε απελευθερώσει και άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για θέματα ενέργεια Και βεβαίω θέλουμε να εμβαθύνουμε το εμπόριο και τι πολιτικέ μα σχέσει. Επίση, το σχέδιο δράση αναφέρει ενδυνάμωση του διαλόγου σε όλα αυτά τα θέματα εν ώψη τη δεύτερη συνόδου κορυφή με το Πακιστάν κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία. Επίση, καθιστούμε σαφέ ότι θα παράσχουμε έμπειρο γνωμοσύνη και για το Αφγανιστάν και για το Πακιστάν και για του ε, γείτονέ του, ε, ιδιαίτερα για την Ινδία. Δεν υπάρχει μαγική λύση για την υπέρβαση των εντάσεων. Πρέπει όμως μη τι άλλο να καταπολεμήσουμε τη δυσπιστία και να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνη. Αυτό καλούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη. Η εφαρμογή των σχεδίων για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι κεντρική σημασία. Είναι μια κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και των θεσμικών οργανών της Ενώσεως. Είναι ένα άνευ προηγουμένο εγχείρημα που αν επιτύχει θα δώσει πολύ <clears throat> εδώ και πολύ καιρό αναμενόμενες λύσεις. Βεβαίως δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ούτε έχουμε μόνο αυτές τις χώρες. Είναι ολόκληρη η περιοχή της ε, Κεντρικής Ασίας που μας απασχολεί. Χρειάζεται λοιπόν αποφασιστικότητα από όλους και συνέπεια μεταξύ των δωρητών και στο ιστορικό των κρατών μελών. δεν θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα αυτά, ούτε αυτές οι χώρες μπορούν ακόμα να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Οπότε ε, χρειάζεται να καλύψουμε, να υπερκεράσουμε τις δυσκολίες που τροφοδοτούν τον ε, εξτρεμισμό και ελπίζω ότι στην προσπάθειά μας αυτή το Κοινοβούλιο θα μας υποστηρίξει. Τώρα το λόγο θα πάρουν οι ομιλητές εκ μέρους των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων. Ο πρώτος, ο κύριος Κασουλίδης, εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για δύο λεπτά, κύριε Κασουλίδη. Κύριε Σκοπός στο Αφγανιστάν της κίνησης ήταν να καταπολεμήσει τους Ταλιμπάν που προσφέρουν καταφύγιο στην Αλκάιδα. Δεν έχει κατανικηθεί η εξέγερση εκεί αποδείχθηκε ότι η νίκη δεν μπορεί να προκύψει μόνο με χρήση στρατιωτικών μέσων. Μόνο με τη στρατιωτική βία και την θανάτωση ε, των εξεγερμένων δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ικανότητα του Αφγανιστάν να ε, εξασφαλίσει την ασφάλειά του, συνεργασία κυρίως στο τοπικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται ενθάρρυνση σε μια διαδικασία συμφιλίωσης στο ίδιο το Αφγανιστάν με αφγανική ηγεσία και καθοδήγηση το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στους μη στρατιωτικούς τομείς. Ωστόσο, εγώ ανέμενα περισσότερη έμφαση για τα θέματα των ναρκωτικών. Το είπατε και εσείς κυρία Υπουργέ και πιο αυστηρές διατυπώσεις και προειδοποίησεις για θέματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Ναι λοιπόν στο ε, σχέδιο δράσης, αλλά διασυνδέονται τα πράγματα αυτά και χρειάζεται επιτυχία και, στους δύο, και στις δύο, στα δύο μέτωπα. Η διπλωματία απαιτείται για να αποφευθεί ώστε το, η σπιστία μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν να, να αποβεί προκόλλημα για την περαιτέρω επιτυχία. Γέρι εκ των Σοσιαλιστών και, και, και Δημοκρατών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρία Υπάτε εκπρόσωπε. Με τη συζήτηση αυτή το Κοινοβούλιο θέλει να συνεισφέρει στην ε, ασφάλεια και σταθερότητα αυτή τη περιφερεια, που είναι ζωτική σημασία για όλο τον πλανήτη. Όλη η νέα στρατηγική που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ομπάμα ε, οδήγησε στην αποστολή νέων στρατευμάτων με πρώτη στο στόχο την προστασία του πληθυσμού και την ενδυνάμωση των ε, δυνάμεων ασφαλείας αλλά και την προστασία των ίδιων των πολιτών. Σωστό είναι αυτό διότι είχε ξεφύγει από τον ελεγχό μας η κατάσταση και προηγουμένως είχε επικεντρωθεί όλη η στρατηγική δύναμη στην καταπολέμηση των Ταλιμπάν. Είναι όμως μια μεταβατική φάση προς ένα Αφγανιστάν ευήμερο και αυτόνομο δημοκρατικό που να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Η βοήθεια λοιπόν της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει ε, και στο πολιτικό και στο μη στρατιωτικό τομέα να επικεντρωθεί μετά από αυτή την πρώτη στρατιωτική φάση. Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, σωστή διακυβέρνηση, καταπολέμηση της διαφθοράς, εθνική συμφιλίωση και σταθεροποίηση της κατάστασης στο Πακιστάν. Εδώ βρίσκεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη έχει ήδη προσφέρει πολλούς πόρους ένα δι στο Αφγανιστάν 300 εκατομμύρια στο Πακιστάν αποστολές πολύ σημαντικές παρά τα προβλήματα προσωπικού η Διεθνής ε, Αποστολή για τις Εκλογές, η Αποστολή Ίζαφ. Παρόλα αυτά, η δυνατότητά μας να επηρεάσουμε τα πράγματα σημαντικά υπολείπεται λόγω οικονομικών ε, προβλημάτων και προβλημάτων ανθρωπίνων πόρων. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε πιο συνεπή την δέσμευσή μας από την πτυχή της πολιτικής και μη στρατιωτικής ενίσχυσης και παρέμβασης. στο σχέδιο δράσης, υπ' αυτή την έννοια, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου. Εμείς το υποστηρίζουμε και ζητούμε την πραγματική του και συγκεκριμένη του εφαρμογή. Συγχρόνως, θεωρούμε ότι οι στόχοι από το σχέδιο δράσης ε, περνούν και από τον εντοπισμό συγκεκριμένων ad hoc μέσων για την ενδυνάμωση των μέσων που έχουν ε, οι το αποστολές. Ε, φόλων αυτών των θεμάτων είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε την υποστήριξή μας. Κύριε Γκουλτιέρη, αλλά ξεπεράσετε πολύ το χρόνο ομιλία σας. Ελπίζω οι επόμενοι ομιλητές να τον σεβαστούν. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Αρλάτσι από την ομάδα των φιλελευθέρων. Thank you. Thank you very much. We are... Ευχαριστώ πολύ. Τι δούμε αυτό το νέο πρόγραμμα δράση για Αφγανιστάν και Πακιστάν. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μου έδωσε την ευκαιρία να αναλάβω την σχετική έκθεση. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική. Χρειαζόμαστε αυτή τη νέα στρατηγική γιατί η μέχρι σήμερα βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν ήταν τόσο συνεκτική, τόσο συνεπής και δεν είχε τόσο σημαντικό αντίκτυπο, κυρία Στον, λυπάμαι. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που μας είπατε στην αρχή για το Αφγανιστάν. λόγο, γραφειοκρατικό ήταν αυτό το οποίο μας είπατε. Ακριβώς όπως και το σημερινό πρόγραμμα δράσης. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει διορθωτικές κινήσεις και να αποκτήσουμε μια πιο αποφασιστική και συνεπή πολιτική. Επί τη βάση των πληροφοριών δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι ακόμα και τα πιο βασικά στοιχεία δεν υπάρχουν για το τι έγινε, τι, τι, τι, τι έχει δαπανηθεί από το 2001. Τι έγινε τα κονδύλια, ποιος είναι Ξέρουμε ότι έχουμε ένα δις ευρώ που έχουν δαπανηθεί εκεί, που είναι πολλά λεφτά. Μιλάμε για 6,9 δις ΑΕΠ της χώρας. Επομένω αυτή η πολιτική αρρωγή είναι το 20% του ετήσιου ΕΠ της χώρας. Επομένως θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τη χώρα να βρει μια καλύτερη τύχη. Επομένως θα πρέπει καταβληθούν κάποιες προσπάθειες να δούμε ποια είναι τα συμφέροντά μας στην ε, περιοχή. Ναι, τελειώνω τώρα. Οπότε εγώ θα ασχοληθώ στην εκθεσή μου και με το πώ θα καταπολεμηθεί η καλλιεργία του όποιου μέσω εναλλακτικών καλλιεργιών. Η κυρία Λάμπερτ για 1,5 λεπτό από την ομάδα των Πρασίνων. Thank um, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένα θέματα με ικανοποιούν στο σχέδιο δράσεως. Άλλοι συναδελφοί μου είπαν ωστόσο ότι ορισμένα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί Το θέμα το εξετάζουμε από την δική μας σκοπιά και καμιά φορά υποτιμούμε την καθημερινή πραγματικότητα και των Αφγανών και των Πακιστανών. Με πολλούς θανάτους, σε βάρος για παράδειγμα των Χαζάρων, με πολλούς φόνους, με ε, επιθέσεις κατά των ε, σχολείων θηλαίων, με επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων κλπ. Η αστυνομική εκεί δεν είναι παρατροφή για τις ε, βόμβες των Ταλιμπάν. δεν έχουμε επιτύχει αυτά που ελπίζαμε πηγαίνοντας εκεί. Χαίρομαι που η Επίτροπος μιλεί για την έναρξη μιας συνεργασίας που θα περιλαμβάνει και την Ινδία. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή και πρέπει να ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις συγκρούσεων όπως το Κασμίρ, όπου ο Αφγανός πρέσβης πριν από λίγες μέρες μας είπε ότι προκαλεί πρόβλημα σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται εκεί. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία και του Πακιστάν πρώτα-πρώτα ε, να εξετάσουμε τι υποστήριξη δίνουμε. Πρώτα-πρώτα στις πολλές χιλιάδες εκτοπισμένων. Και η έλλειψη εμπλοκής μας με τους εκτοπισμένους στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν στο παρελθόν που έχει αφήσει ένα κενό. Και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση, στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και βεβαίως ιδίως των εκτοπισμένων. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη στρατιωτική αποστολή ΝΑΤΟ-ΑΕΣΑΦ να αποτύχει. Χρειάζεται πολιτική βούληση, εξοπλισμός και μεγαλύτερος αριθμός στρατιωτικών δυνάμεων επιτόπου. Τότε το ΝΑΤΟ μπορεί να νικήσει τους Ταλιμπάν και βέβαια πρέπει ταυτόχρονα να κερδίσει τις καρδιές των ε, ντόπιων. Μέχρι τώρα δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Τώρα υπάρχει και το Ιράν με πυρηνικέ φιλοδοξίες με το Πακιστάν, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το ενισχύσουμε το Πακιστάν. Για παράδειγμα, μέλη της ε, Ιρανικής ε, Υπηρεσίας ε, Πληροφοριών φαίνεται μέχρι τώρα να δίνουν υποστήριξη στους Ταλιμπάν και τώρα μόλις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τους εσωτερικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος που προκαλείται από το Πακιστάν με, την, με το καταφύγιο που δίνει σε τρομοκράτες σε βάρος της Ινδίας αρχίζει και γίνεται κίνδυνος και απειλή για ολόκληρη την περιοχή. Δίνεται υποστήριξη για την καταπολέμηση των τζιχάντης και οικονομική υποστήριξη. Πρέπει ωστόσο να δώσει εγγύησει ότι οι αλλαγές που θα γίνουν εκεί δεν θα οδηγήσουν στην ε, ενίσχυση των συμβατικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ινδία. Τέλος, Αφγανιστάν και Πακιστάν. δεν συμβαδίζουν με την ε, μετριοπαθή στάση της Ινδίας μέχρι τώρα από την Αριστερά για ένα λεπτό Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Η ομάδα μου ποτέ δεν συμμερίστηκε τη στρατηγική του πρώην Πρόεδρου Μπούς στο Αφγανιστάν και ο χρόνος μας δικαίωσε. Αυτή τη στιγμή στο Αφγανιστάν υπάρχει μια νόμιμη μεν διεφθαρμένη δε κυβέρνηση ε, με, πολλά, με πολύ μεγάλες παρενέργειες, με πολλά θύματα. Η κατάσταση των γυναικών δεν βελτιώθηκε καθόλου και λυπούμαστε που και ο πρόεδρος Ομπάμα στέλνει 30.000 ε, ε, περισσότερους στρατιώτες και φαίνεται να σπάζεται την ίδια προσέγγιση. Δεν θέλουμε ένα νέο Βιετνάμ τον 21ο αιώνα. Στο Αφγανιστάν έχει αποδειχτεί ότι η λύση δεν μπορεί ποτέ να είναι στρατιωτική η συνεργασία, η διπλωματία και η συμφιλίωση στην γεωστρατηγική αυτή ζώνη είναι η λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μέγερ, τώρα για ένα λεπτό επίσης η κυρία Σανκλέρ. Thank you, Madam uh, Chairman. Um, I had the pleasure... Είχα την ε, ευκαιρία να συναντήσω κάποιο από τι δυνάμει τη χώρα μα που γύρισαν από εκεί και όλοι μου είπαν το ίδιο. Δεν είναι άρτια εξοπλισμένοι. 40.000 λίρε τη μέρα πληρώνονται σε ένα καθεστώ διεφθαρμένο. Άρα θα έπρεπε να δούμε πώ θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, πώ θα γίνει καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού εκεί. Γιατί πρόκειται για την πιο καυτή, την πιο κρίσιμη, την πιο δύσκολη περιοχή στον κόσμο και άρα εκεί θα πρέπει να σημειώσουμε κάποια βήματα Το πρόβλημά μου είναι ότι μια που δεν έχει πείρα η υψηλή ε, εκπρόσωπος έχουμε πρόβλημα και στην ε, πολιτική μας δεν είχε καμία σχέση με τον κλάδο των εξωτερικών ούτε καν σε, υπουργείο, σε γραφείο ταξιδιών δεν έχει δουλέψει άρα θα πρέπει να παρατηθεί και να αντικαταστήσει άλλος ε, Μπρονς, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, τα συμπεράσματα φαίνονται πάρα πολύ θετικά σε σχέση με την φρύπολη στάση είπα και Ενωμένο Βασίλειο με καλύτερα, που φαίνεται μάλλον αφελή, ίσως και ένοχα. Και το Συμβούλιο επομένω αφελώς θέλει στο εχθρικό έδαφος ε, των φυλών αυτών να μεταλαμπαδεύσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει διαφθορά, λέει το κείμενο. Δεν είναι δυνατόν εκεί ο δικός μας τρόπος ε, δημοσιονομικής διαχείρισης να πιάσει τόπο. Όχι επειδή στα γονιδιά τους έχουν ε, το να είναι ανέντιμη, αλλά επειδή είναι τέτοια δόμη της κοινωνίας και των φυλών. Είπαμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει για το όπιο, είπαμε όμως από την άλλη μεριά ότι δεν απέδωσε και το να φύγουν οι Ταλιμπάν από την κυβέρνηση. Έγινε μείωση 90% όμως από τότε που έγινε η εισβολή και μετά ξαναγίνανε η πιο σημαντική παραγωγή του οποίου λέει επίση στο κείμενο επιλέξει ότι η ανασφάλεια δεν είναι να αντιμετωπιστεί μόνο με στατικά μέσα τέλο τη παράθεση. και αυτό όμω τι σημαίνει ότι θα πρέπει κάτι να γίνει με, μέσω της πολιτικής οδού της δημοτικής οδού Είχαμε όμως ε, τρεις αποτυχημένες επεμβάσεις εκεί, 19ο αιώνα, καταπιέζονται και οι γυναίκε, υπάρχει περιφέρεια για τη δημοκρατία, σκοτώνονται οι στρατιώτες μας ε, πάρα πολύ δυσάρεστο όμως, μπορούμε να το σταματήσουμε αύριο. Πώς, εάν μετακαλέσουμε εδώ, εκεί, τις δυνάμεις μας. Αυτόν τον πόλεμο δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε. Η διεθνή κοινότητα και όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν πρόβλημα στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος Ομπάμα πήρε τρεις μήνες μέχρι να αποφασίσει μια στρατηγική για να ε, δώσει μια απάντηση στην ανησυχητική έκθεση του στρατηγού Μακρίσταλ. Βραχυπρόθεσμη αναδίπλωση στρατευμάτων, σταδιακή μεταφορά προς τις ε, αφγανικές δυνάμεις, καλύτερο συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και καθορισμός πολιτικών προτεραιοτήτων. Τώρα, κυρία Άστον, η πρόκληση είναι η ευρωπαϊκή απόκριση μέσω της διασκέψεως του Λονδίνου. Εσείς στην ε, παρέμβασή σας αναφέρατε δύο λέξεις κλειδιά. Μια απόκριση, είπατε, συντονισμένη με τα άλλα διεθνή βήματα και αυτό το υποστηρίζουμε. Και μια απόκριση, είπατε, συνεπή Επ' αυτού δύο σχόλια. Το 2005 είχα το προνόμιο να είμαι επικεφαλής μια αποστολής αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με τον ε, στρατηγό Γκρατσιάνο. Έχουμε μια πολύ ετηρογενή στρατιωτική παρασία που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. Το δεύτερο κυριάστον είναι ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο στο Αφγανιστάν γιατί περί πολέμου πρόκειται χωρίς να έχουμε μαζί μας τον εντόπιο πληθυσμό. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό. Ένα δις ευρώ που έχουμε δαπανίσει να δαπανίσουμε για να κερδίσουμε τον λαό. Θα ήθελα να θυμηθώ τρολογία 23 ετών που προερχόταν από την εκλογική μου περιφέρεια και πέθανε στην επαρχία Πρόβενς στις 7 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι σκέψεις μας να στραφούν στην οικογένειά του και σε όλες τις οικογένειες ευρωπαϊκές, αφγανικές και πακιστανικές που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Μπροστά σε τέτοιε θυσίες καθήκον δικό μα είναι να φροντίσουμε να πράξουμε πάντα το δυνατό για να προαγάγουμε την ειρήνη και την ευημερία στο Αφγανιστάν. Εάν θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τι απαραίτητε αλλαγέ και στην ε, κοινή εξωτερική πολιτική, το πρώτο μέρος όπου έπρεπε να δράσουμε είναι το Αφγανιστάν. Να φροντίσουμε ώστε να συντονιστούν οι δραστηριότητες των χωρών μελών και να ταχθούν όλες πίσω από αυτή τη νέα στρατηγική. Χαίρομαι για τη δέσμευση της, υπά, της εκπροσώπου για την μετάβασή της επιτόπου στο νέο έτος, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και την ίστατη δοκιμασία για ε, την ε, πολιτική αυτή. Τέλος, οι χώρες μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ώστε η Ιούπολ να δώσει τους ε, αξιωματούχους που έχει υποσχεθεί για να εκπαιδεύσουν τους Αφγανούς αστυνομικούς ώστε να μπορούν αυτοί να τα αποκριθούν στα καθήκοντά τους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να σας τονίσω ότι είμαι κατά των όσων είπε η κυρία Σενκλέρ, κατά της κυριά Άστον πριν από λίγα λεπτά πρόεδρε, στο Αφγανιστάν. Ένα παιδί στα τέσσερα δεν φτάνει στην ηλικία των πέντε ετών. Αυτό στο δημοκρατικό έλλειμμα έχουμε έλλειμμα και στην ασφάλεια και στις συνθήκες ε, υγείας. Οπότε ε, έχουμε ευξήμενη κινητικότητα των Ταλιμπάν και επομένως χρειάζεται κάτι να γίνει όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση του προβλήματος του Αφγανιστάν μόνο με στρατιωτικά μέσα δεν γίνεται τίποτα. Παρά το ότι έχουμε πολλά με τη διάθεσή μα. Και όσον αφορά τη ε, στρατιωτική πτέρυγα των δυνάμεων εκεί, είναι υπεύθυνο το να το οποίο μα είδε ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων του. Ανθρωπιστική βοήθεια, συνεργασία αναπτυξιακή, όλα αυτά δεν είναι συνταγή δοκιμασμένη. Όμω χωρί ε, αυτά δεν θα πετύχει το ΝΑΤΟ. Επομένως χρειάζεται να βρούμε για τους Αφγανού κάποιες προοπτικέ πιο ευίωνε. Η ευθύνη μας είναι βαριά. Στο Αφγανιστάν ακόμα είναι ο λαό διχασμένο. το κράτος ανοργάνωτα. Μην ξεχνούμε ότι οι περισσότεροι Αφγανοί θέλουν την ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι το εργοσυσήφιο, αλλά δεν μπορούμε εμεί να σταυρούμε τα χέρια για να αφήσουμε αυτή τη χώρα να είναι θύματα των, των φανατικών. Νίλσεν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Merci. Ευχαριστώ. Ναι, πρέπει να βγούμε από την παγίδα στην οποία πέσαμε με την πολιτική Μπούς. Όχι πότε, πώς θα πρέπει να αποχωρήσουμε, πρέπει να αποφασίσουμε. Αλλιώς θα χάσουμε πλήρως την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του αφγανικού λαού και θα την κερδίσουν οι Ταλιμπάν. Η στρατικοποίηση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να πάυσει, διότι δημιουργεί σύγχυση ε, και καθιστά τις ε, ΜΚΟ αναξιόπιστες. Πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στην αναφιόμενη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, στους ρεφορμιστές και μεταρρυθμιστές. Γιατί δράτουμε έτσι, γιατί βοηθάμε το Αφγανιστάν, γιατί το αποφάσισαν οι Αμερικανοί ή για να το βγάλουμε από τον σκοταδισμό θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στις υπηρεσίες προς το λαό, παιδεία, υγεία, μεταφορές, να υποστηρίξουμε την τοπική διαχείριση και διακυβέρνηση. Η κουλτούρα αυτής της χώρας δεν είναι ίδια με τη δικιά μας. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κυρία Μπίμπα Σάραμπη, η κυβερνήτη της Μπανιάρ, πρώτη γυναίκα κυβερνήτη. Πήγαμε το 2001, θα θυμάστε, επί τόπου για να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Βανόρντεν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Uh, Madam President, uh, to read the EU Action Plan for Afghanistan and Pakistan. αυτό το πρόγραμμα δράσης και μπορούμε να φανταστεί κανείς πώς είναι η κατάσταση. Όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνουμε εμείς. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να γίνει διαφορά, όμως θα πρέπει αυτά να γίνουν στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας διεθνούς κοινότητας και εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία την προσπάθειά μας, ώστε να μπορέσουμε ε, κάτι να κάνουμε. Ε, το δικαίωμα είναι πάρα πολύ σοβατικό. Πάντως, σε αυτές τις 12 σελίδες βρίσκω μόνο τέσσερις αναφορές της ε, ΕΠΑ και μόνο μία στο ΝΑΤΟ. Όμως, αυτοί οι παράγοντες είναι η εγγύηση της επιτυχίας, γιατί αν δεν υπάρχει ασφάλεια και σταθερότητα δεν είναι τον έχουμε χρηστεί διακυβέρνηση κανένας είδους ε, πρόγραμμα συγκέντρωσης που να έχει νόημα ούτε ανάπτυξη. Όσο αφορά τώρα τα πολιτικά μη στρατικά μέσα. Έχουμε δώσει τόσα δις από το 2001. Τεράστιο το ποσό που έχει δαπανηθεί, όμως δεν υπάρχει, δεν έχουμε κάνει τη διαφορά. Άρα δεν έγινε διασπάθηση. Επομένως χρειάζεται μια σφαιρική προσπάθεια, διεθνής προσπάθεια για Αφγανιστάν και Πακιστάν. Ακόμα όμως δεν μπορώ να δω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συμπλέψει με τη διεθνή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οκτώ χρόνια μετά γνωρίζουμε όλοι ότι η μέχρι τώρα στρατηγική στο Αφγανιστάν που βασίζεται στο, στη στρατιωτική δράση έχει αποτύχει. Αφενός λοιπόν έμφαση στο στρατιωτικό, αφετέρου περιορισμένη πόροι για, τη, για, τους, για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες των πολιτών. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή της στρατηγικής. Να ξεφύγουμε από τη στρατηγική δράση και να πλησιάσουμε τους ανθρώπους. 40% των Αφγανών είναι άνεργοι. Περισσότεροι από τους μισούς Αφγανούς ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Μπορούμε να τους προσφέρουμε εκπαίδευση. Μπορούμε να θέσουμε το κοινωνικό θέμα στο επίκεντρο. Αυτά αναμένουμε από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως, χρειάζεται και η ενίσχυση της υπεύθυνη κυβέρνησης Χρειάζεται συμμετοχή των Ταλιμπάν. Όποιος όμως κινείται μόνο μέχρι τα μισά του δρόμου και συνεχίζει να προχωρεί σε στρατιωτικές περιπέτειες, χάνει το τρένο τελικά και είμαστε στο 12 παρα 5. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτές τις ε, πολύ περίπλοκες και δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε απλές ιδέες. Η πρώτη απλή ερώτηση είναι γιατί πήγαμε στο Αφγανιστάν. Με ένα στόχο να καταστρέψουμε τα στρατόπεδα εκπαίδευσης των Ταλιμπάν, εφαλτήριο για την διεθνή τρομοκρατία που μας απειλούσαν. Σήμερα δεν υπάρχουν. Δεύτερη παρατήρηση. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δυστυχώς οι στρατιώτες θεωρούνται, οι στρατιώτες ε, της ε, Δύσης θεωρούνται ε, κατακτητής και όχι α, φίλος. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όποιοι διαδίνονται το αντίθετο, τους καλούν να πάνε εκεί να δουν τι γίνεται επί τόπου. Τρίτο, η κατάσταση από ασφάλειας είναι πολύ επιδεινωμένη. Το 2004 μπορούσε κανείς να περπατήσει στην Καμπούλ, σήμερα αυτό είναι αδύνατο. να εφαρμόζουμε ακόμα παλαιές μεθόδους και να μην ε, ε, διδασκόμεθα από τα λάθη μας είναι θελοτυφλία. Οι συνέπειες. Διαλύσαμε τα στρατόπεδα της Αλκάιντα και πρέπει να αποχωρήσουμε. Μπορούμε να αποχωρήσουμε τώρα. Όχι. Γιατί αυτό θα δημιουργούσε χάος και επιστροφή των στρατοπέδων. Πρέπει να αποχωρήσουμε υπό προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η αυγανοποίηση, να δώσουμε τα κλειδιά της λύσης στους ίδιους τους Αυγανούς. Το δεύτερο είναι, και το συζητήσαμε αυτό με όλους τους, ε, να συζητήσουμε με όλες τις δυνάμεις, με όλους τους διαφωνούντες, ε, τους εξεγερθέντες και να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι τα ευρωπαϊκά κριτήρια αυτά που θα προτανεύσουν ούτως ή άλλως στο Αφγανιστάν δεν είναι η ίδια η κοινωνία, δεν έχει οι ίδιες παραδόσεις, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, διότι τελείως θα αποτύχουμε και μάλιστα παταγωδός. Ευχαριστώ κύριε Ζιβάν. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Το Συμβούλιο λέει ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη. Όντως, αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να δώσουμε προς τους Ευρωπαίους πολίτες με ειλικρίνεια και θάρρος Υπό αυτή την έννοια χαιρετίζω το νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πακιστάν και το Αφγανιστάν που προβλέπει ένα τεράστιο πρόγραμμα capacity building για τις δύο χώρες. Μόνο με την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσεως ως διαμεσολάβηση της Ευρώπης μπορεί να οικοδομήσουμε δομές και θεσμούς που θα βάλουν τέρμα στον πόλεμα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τους Αφγανούς και δεν είμαστε εκεί επειδή το αποφάσισαν οι Αμερικανοί. Η παρουσία μας θα είναι ε, απαραίτητη για πολλά περισσότερα χρόνια και όχι μόνο στρατιωτική και μη στρατιωτική. Τώρα, η... καταγγέλλω την ε, διαβίας επιστροφή, αναγκαστική επιστροφή Αφγανών πολιτών στο Αφγανιστάν. Από τη γαλλική κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα πράγμα που δεν χρειάζεται στην πικρή αυτή πραγματικότητα του Αφγανιστάν είναι τα ωραία λόγια. Και απευθύνομαι σε εσά, Λέδη Άστον. Είπατε ότι οι χώρες μέλη είναι δεσμευμένες και ειλικρινά για την ε, εκπαιδευτική αποστολή της UPOL. Το βλέπετε πραγματικά αυτό και ούτε καν καταφέρνουμε να συνάξουμε τους 400 αστυνομικούς. Πρόκειται για διγλωσία και γελιότητα. Εάν είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε, τότε πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Ήδη προδιετίας το European Security Review διεπίστωνε ότι ο μικρό αριθμός αστυνομικών εκπαιδευτών στην ουσία αμφισβητεί την δέσμευση της Ευρώπης. Γιατί δεν χρηματοδοτούμε εκπαιδευμένου αστυνομικού εκεί στο Αφγανιστάν αρκετά ώστε να αποτρέψουμε να πάνε στους Ταλιμπάν. Θα μας κοστίσει λίγα χρήματα και θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα. Η Ευρώπη, λέει Άστον, λέει πολλά και μεγάλα λόγια. Είναι ντροπή όμως το πόσο μικρά και ντροπαλά τα έργα της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστά λέγεται νέα δράση για Αφγανιστάν και Πακιστάν. Αυτά όμως που λέχθηκαν στο πλαίσιο αυτό μου φαίνεται σαν να είναι περισσότερο δύο ξεχωριστά σχέδια δράσης τα οποία παρουσιάστηκαν το ένα μετά το άλλο. Κάτι λέχθηκε για τις δύο χώρες. Εγώ θεωρώ ότι στο Αφγανιστάν ε, πρέπει να έχουμε μάθει κάτι από τα <clears throat> σφάλματα του παρελθόντος και θα κάνουμε προσαρμογή των πολιτικών μας και των δομών μας. Για το Πακιστάν χαίρομαι που η νέα πολιτική θα ακολουθήσει την έκθεση της παρατήρησης εκλογών στην οποία, την οποία θα συντάξει εγώ. Και οι συστάσεις αυτές της, αυτής της έκθεσης θα <coughs> μεταφερθούν στην πραγματική καθημερινή πολιτική. Ωστόσο, ελπίζω στη δευτερολογία τους το Συμβούλιο και η Κομισιόν να δηλώσουν ποια θα είναι η κοινή στρατηγική για τις δύο αυτές χώρες. Διότι διαπιστώνουμε ότι οι χώρες αυτές μοιράζονται ένα σύνορο χιλιάδων χιλιόμετρων που δεν μπορεί να ελέγχεται από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά οι πολιτικές που ασκούμε είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά έχουν άμεσες συνέπειες και πέραν των σύνορων αυτών. Ποιες Δομέ λοιπόν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε εκεί. Πώς θέλουμε να κινηθεί ο διάλογος μεταξύ πακιστανική και αφγανική κυβερνήσεω. Πώ Θέλουμε να αναπτύξουν νοοτροπία οι άνθρωποι εκεί επιτόπου ώστε να αποδεχθούν τις πολιτικές αυτές. Σε αυτά τα ερωτήματα χρειαζόμαστε απαντήσεις και ελπίζω να τις λάβουμε. Λόγω τώρα ο κύριος Πάσχου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank you, Madam President. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το πρόγραμμα δράση για Αφγανιστάν και Πακιστάν που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο, καταρχήν είναι αξιόλογο. Αντιστροφή τη ευθύνη, λέει. Δηλαδή να περάσει την εθνική κοινότητα στο αφγανικό κράτο και εμεί να έχουμε ρόλο υποστήριξη. Και όσον αφορά του επιπλέον 3.000 άντρε, είπαμε ότι μέχρι το 2011 θα αρχίσει τότε η απόσταση των ΗΠΑ και θα περάσει η ευθύνη στο Αφγανικό κράτος. Έχουμε τους ίδιους στόχους με τι ΗΠΑ. Δηλαδή πώ θα αναλάβει τα ενία τη κατάσταση ε, το Αφγανικό κράτος όμως. Το χρονικό πλαίσιο μεταξύ ημών και εκείνων διαφέρει. Θα πρέπει μέχρι το 2011 να έχουμε πετύχει έναν σημαντικό βαθμό ασφάλειας. Όμως η σταθερότητα θα παργήσει περισσότερο. Επαρκής ε, ασφάλεια δεν θα έχει εξαφανιστεί το 2011 και όταν φύγουν οι Αμερικανοί τα πράγματα θα χειροτερέψουν οπότε μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ασφάλεια τότε αν όχι τότε έχουν πρόβλημα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαιρετίζουμε με το γεγονό ότι η Σουηδική Προεδρία θέλει να βοηθήσει να αναβαθμιστεί ο ρόλο μα όσον αφορά το Αφγανιστάν. Όμως το θέμα τι θα γίνει με την χρηματοδότηση αυτού του πρόγραμματο δράση. γιατί από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ σημαντικός σταθμό θα είναι η διάσκεψη του Λονδίνου του Ιανουαρίου. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τη νέα κυβέρνηση τη χώρα. Θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ε, διαφθορά, τι θα γίνει με τα ναρκωτικά και με ανησυχούν αυτά που γράφει σήμερα ο τύπο όσον αφορά τη διάσκεψη που προείδρευσε ο Καρζάη όσον αφορά την διαφθορά. Επίση, ο πρώτο Ομπάμα είπε ότι θα πάει στι 30.000 στρατιώτε. Όμω, η χώρα ζει κρίσιμε στιγμέ. Επομένω, θα πρέπει οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι να συντονίσουμε τις προσπαθίε μα. Γιατί αυτό το οποίο διακυβεύεται εκεί δεν είναι μόνο η ευημερία και η ελευθερία των Αφγανών, αλλά η σταθερότητα σε ευρύτερη το, κάτι το οποίο αγγίζει για μια τόσο σημαντική χώρα στο Πακιστάν επίσης είναι και θέμα δικής μας ασφάλειας διότι συνεχίζει η, η σκιά της απειλής της τρομοκρατίας άρα το τι θα πετύχουμε στο Αφγανιστάν θα εξασφαλίσει το τι θα γίνει στην Δύση δεν είναι δυνατόν να αποτύχουμε αλλά χρειαζόμαστε στήριξη από τους Ευρωπαίους για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να είναι ξεκάθαρα, κρυστάλλινα, διάφορα τα πράγματα θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος όσοι πάνε στο Αφγανιστάν πόσο κινδυνεύουν, αλλά επίση θα πρέπει και να σταθούμε στο πόσο σημαντική υπόθεση είναι το τι κάνουμε στη χώρα αυτή και το ότι δεν επιτρέπεται να αποτύχουμε. Πάρα πολλά διακυβεύονται. Ένας Αφγανός φίλος μου είπε κάποτε ότι είναι καλό που μπήκε η Δύση στο Αφγανιστάν μη λησμονείτε όμως ότι κάθε εισβολέας που μπήκε στο Αφγανιστάν για παραπάνω από ένα χρόνο έμεινε εκεί πάρα πολύ. Το 2001 είχαν γίνει αυτά, τώρα είμαστε το 2009. Πρέπει να δούμε ότι ποια είναι η στατιστική πορεία μέχρι τώρα. Οι λένε ότι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα στρατιωτικά. Μια τέτοια χώρα ποτέ δεν διοικήθηκε κεντρικά. Πώς θα την κάνουμε τώρα. Δηλαδή θα ρίξουμε όλο το βάρος μας στην κατανίκη της Αλκάιντα και μετά θα φύγουμε. Πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αυτό. Καθώς και το ερώτημα του κ. Βανόρντεν σε σχέση με την διαδικτύωση του σχεδίου δράσεως με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους, με το σχέδιο Ομπάμα και ούτω καθεξής. Είναι σωστά αυτά. Και σωστά να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των περιπτώσεων Πακιστάν και Αφγανιστάν και βεβαίω συμφωνώ και με όσα λέχθηκαν για τι Ινδίε. Και τέλο πρέπει να δούμε πώ εξελίσσεται εσωτερικά η χώρα αυτή. Μέχρι τώρα ποτέ δεν έχω δει όταν ασκείται στρατιωτική πίεση εκ των έξω και έχουν εκπαιδευτεί στρατιωτικοί και αστυνομικοί που δεν έχουν όμως ξεκάθαρο στόχο. Δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει ιδεολογική υποστήριξη μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο όπου τελικά ποτέ δεν κερδίζουμε. Γι' αυτό φοβούμε λοιπόν ότι είναι κατακαιρματισμένες οι προσπάθειές μας και ίσως πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε με ποιο σχέδιο πράγματι μπορούμε να κάνουμε να, ε, να αποσύρουμε τις θετικές μας δυνάμεις από εκεί, ταυτόχρονα σταματώντας την τρομοκρατία. Στη διαδικασία Catch the Eye έχουν ζητήσει το λόγο αρκετοί συνάδελφοι. Ε, σας παρακαλώ μην ξεπερνάτε το ένα λεπτό για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο δυνατόν περισσότερο. Ξεκινάμε με την κυρία Κόμη. Η κυρία Κόμη. Η ασφάλεια στο Αφγανιστάν ε, υπέστη πρόσφατα μεγάλη επιδείνωση λόγω της έλλειψης ε, ελέγχου της επικράτειας ε, από τις ε, φυλές διοικούνται ευρύτατες περιοχές της χώρας και κομμάτια των πόλεων παρά την ε, παρουσία των δυνάμεων της ISAF. Η τρομοκρατία συνδέεται άμεσα με αυτό και γι' αυτό είναι απαραίτητο να παραμείνουν η ΕΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχες χώρες. Αυτό είναι προφανές. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε μόνο με στρατιωτικά μέσα να αντιμετωπίσουμε την κρίση και για το Αφγανιστάν και για το Πακιστάν. Το νέο σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί από αυτή την έννοια ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση τη ασφάλεια στα πλαίσια τη ε, ευάλωτη διαδικασία του capacity building, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ε, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Παρακαλώ, κύριο za zabranie głosu. Otóż ja uważam, że plan Unii Europejskiej... Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ισορροπημένο, είναι σωστό, γιατί μια τέτοια ενίσχυση πρώτη χώρα θα πρέπει να στεφτεί και από δύο άξονε πρώτα πρώτα την ασφάλεια και δεύτερον ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου τη χώρα. Όσον αφορά την ασφάλεια, τώρα, εάν τα πάμε καλά, τότε συνακόλουθα θα προτείνει και το βιωτικό επίπεδο. Και εάν ανέβει το βιωτικό επίπεδο, αντιστρόφως πρόκειται και η ασφάλεια να αναβαθμιστεί. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει η αρρωγή μας προς αυτή τη χώρα να είναι αποτελεσματική και για να είναι πιο αποτελεσματική θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη των χρόνων της Κεντρικής Ασίας. Επομένως, κυρία Άστον και κυρία Μάλμστρομ, θα πρέπει να συνεχίσετε τι επαφέ σα με το Τατζικιστάν. Είναι μια χώρα που μπορεί να μα βοηθήσει στο στόχο μα. Θα βοηθήσουν από την επιμελητία και τι μεταφορέ. Οι, βόμβες βάζουν, οι τρομοκράτες βάζουν καθημερινά βόμβες σε σχολεία, σε ε, καταστήματα ακόμα και σε στρατιωτικά επιτελεία. Οι πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποκρούν τους Αφγανούς που ε, προσπαθούν να διέρθουν τα σύνορα. Όμως οι τρομοκράτες αυτοί από πού βρίσκουν όπλα είναι υπεραπλουστευτικό να πούμε ότι είναι εσωτερικό θέμα του Πακιστάν. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Η Υπουργό κ. Μάλμστρομ σωστά έθεσε το θέμα της περιφερειακής πολιτικής με το νέο ρόλο της είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Θα ενισχύσουμε τους Πακιστανές να κάνουν ό,τι μπορούν. Και ταυτόχρονα είναι σωστό ότι ναι μεν υπάρχει αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ Πακιστάν και Ινδιών και εγώ με ασφαλώς υπέρ της συνεργασίας των δύο αυτών χωρών διότι όσο εξακολουθεί η δυσπιστία αυτή πολύ μικρή πρόοδος μπορεί να γίνει. Και όσο το κεντρικό θέμα του Κασμίρ εξακολουθεί να υπάρχει, φοβούμαι ότι δεν θα κάνουμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω το πρόγραμμα για το Αφγανιστάν ε, είναι ένα μεστό, λογικό πρόγραμμα αλλά ίσως ε, υπερτονίζει τον δικό μας ευρωπαϊκό ρόλο. Είμαστε δεσμευμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση, αλλά θα πρέπει να δούμε και οι σύμμαχοί μας τι θέλουν να κάνουν. Αυτό το πρόγραμμα δράση θα πρέπει καταρχήν να ποντάρει στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών σε μη στρατιωτικά μέσα παρέμβασης ε, θα πρέπει να παραιτηθούμε από την ιδέα της κυριάρχησης ε, στο Αφγανιστάν με στρατηγικά μέσα, μια που δεν έχουμε την υποστήριξη του, του, του λαού, γιατί οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να θεωρούνται ως λαϊκή, λαϊκό ένοπλο, ένοπλο κίνημα. Άρα θα πρέπει να βρούμε μια περιφερειακή λύση και έτσι οι γείτονες του Αφγανιστάν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά λέξαν για το σχέδιο δράση για το Αφγανιστάν. Λυπούμε προσωπικά που από τι παρουσιάσει που έγιναν σήμερα δεν ε, τέθηκε περισσότερη έμφαση στην διασύνδεση τη ε, ΕΟΠΟΛ με την ε, αποστολή του ΝΑΤΟ και ποσοτικά και ποιοτικά τα προβλήματα που έχουμε ε, είναι λόγω έλλειψη συντονισμού, αποτελεσματικού συντονισμού. Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, ξέρουμε ότι χρόνια στάθεια αποτολεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα όχι μόνο για τη χώρα, αλλά την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Αφγανιστάν. Ε, στο Πακιστάν υπάρχει μεγάλη ιδεολογική εγκύτητα και πολλές φορές ε, και πρακτική εγκύτητα ε, μεταξύ εξτρεμιστών του Κασμίρ και, που δρούν και στην ε, Μεθόριο ε, με το Αφγανιστάν. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα έχουμε υπόψη μας για να μην δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις εγκύτητες να έχουν καταστροφικές παρενέργειες. Ποιος Κόρτες έχει το λόγο τώρα. Κόρτες Λάστρα. Λοιπόν, η κυρία Κρέσου έχει το λόγο. Η χώρα αυτή μαστίζεται από αυτού του πολέμου που προηγηθεί. και είχαμε δύο ε, αυτοκρατορίε, πρώτα τη Βρετανική και κατόπιν την Σοβιετική, που επέπεσαν στη χώρα. Όμω δυστυχώ τελικά οι Ταλιμπάν κύραξαν στη χώρα, οπότε οι γυναίκε έχουν σε δυσμενή θέση, φτώχεια, ναρκωτικά και όλα αυτά ε, έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ το έργο μας. Επομένως θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή τη βία, σε αυτό το χάος που κυριαρχεί στη χώρα και να δούμε πώς και η στρατιωτική μα αποστολή εκεί θα είναι πιο αποτελεσματική και πώ επίση θα βοηθήσουμε τον εξονισμό και τον οργανισμό τη χώρα. Χρειάζεται επομένω ε, μία αρρωγή προς τη χώρα αυτή, δηλαδή να καταλάβουμε ότι έτσι θα κάνουμε επένδυση για τη δική μας ασφάλεια. Και έτσι πρέπει να μπορέσουμε να γίνει ξανά με φυσιολογική αυτή η χώρα και να αποκτήσουν και ασφαλή πολίτες. Szanowny Panie Przewodniczący, e, sytuacja w Afganistanie jest Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο ε, Αφγανιστάν είναι το πιο οξύ πρόβλημα ε, στην ε, διεθνή σκηνή ιδιαίτερα τώρα μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Η στρατιωτική μας παρουσία ήταν φιλόδοξη αλλά δεν έχει επιτύχει πλήρως. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία μας με την Ινδία, όπως επίσης και στις προσπάθειες ε, ε, για την δημιουργία μιας ε, οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η χώρα δεν έχει παράδοση στον ε, τομέα αυτό. Αυξάνονται πολύ τα, ο αριθμός των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό είναι πολύ ευτυχές και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για την ενδυνάμωση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Äh, vielleicht lassen Sie mich als Mitglied der Iran-Delegation noch eine kurze Anmerkung. machen. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Όταν συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια με τον Ιρανό πρεσβευτή στις Βρυξέλλες γιατί επιβάλλεται θανατικές, επιβάλλονται θανατικές ποινές ε, τέσσερις φορές περισσότερο από τότε που ανέλαβε ε, τα καθήκοντά του ο νέος ε, πρόεδρος. Ε, λάβαμε απάντηση ότι η διαφθορά είναι τέτοια που αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Το Συμβούλιο ευχαριστεί για το τόσο έντονο ενδιαφέρον που πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Κασουλίδη, πρώτα απ' όλα απαντήσω στη δική σα ερώτηση. Το πρόγραμμα δράση λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή πτυχή του θέματο που είναι τόσο σημαντική. Επίση, θεωρούμε ότι όντω η χρηστή διακυβέρνηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να τολμηθεί η διαφθορά και να κυριαρχήσει το κράτο δικαίου. Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν χρειάζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό τη βοήθειά μα και έχει δει ο κ. Κασουλίδη ότι ακόμα δεν μπορούσαμε να κάνουμε αρκετά για το θέμα. Για το θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών. Έχουμε ήδη καταβάλει κάποιε προσπάθειε. υπάρχει τεχνική αρρωγή ω προ όλα αυτά, όμω θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπαθειές μα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ οι προσπάθειες κυβέρνηση τη χώρα αυτής θα ε, στηριχτούν τόσο ώστε να υπάρχει ευημερία και ασφάλεια στη χώρα. Και επίση συμφωνώ ότι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν έχουν περάσει μέσα από έναν σοβαρό συντονισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε γι' αυτό και θα ωφελήσει το παρόν πρόγραμμα δράσης η Ειδική Προεδρία. Πάσχησε κατά την περίοδο του φθινοπόρου το ώστε να εξεύρει το ποιο θα κάνει τι. Οπότε πλέον ξέρουμε το τοπίο καλύτερα. Έχουμε και την έκθεση του Κοινοβουλίου. Συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή σας Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Ντονζό. Εγώ να σας πω ότι η Ιούπολ είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συνεργασία στην περιοχή και ο ρόλος της αστυνομίας επίσης είναι κρίσιμος. Είπαμε ότι χρειάζεται στιβαρή διακυβέρνηση. Νομίζω ότι η συμβολή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάντως δεν έχουμε μπορέσει μέχρι σήμερα για την Ιουπόλ να βρούμε το προσωπικό το παραπάνω που χρειάζεται. Πρέπει να μας βοηθήσουν τα κρατημέλη. Σε έξι στρατηγικά σημεία πρόκειται να ασκήσει τη δράση της Ιουπόλ σε έξι, σε τομείς μάλλον, σε, σε έρευνα, στη ιεραρχία, σε σύνδεση με την εισαγγελία, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφθορά, σε όλα αυτά θα βοηθήσει η αστυνομία μας. Το δε έχει υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Εν κατακλείδη. Πρόεδρε, το πρόγραμμα δράση είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιοποιήσει του πόρου τη αλλά πρέπει να γίνει αυτόν περισσότερο συντονισμό και συνεργασία και θα πρέπει επομένω να εστιάσουμε προσπαθίε μα στην υλοποίηση όλων αυτών των σωστών προτάσεων και να δούμε πώ θα λάβει υπόψη την περιφερειακή διάσταση και να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, και οι αρχές του Πακιστάν και του Αφγανιστάν. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτο δικαίου να είναι στο επίκεντρο αυτή τη προσπάθεια. Πάντως δεν είμαστε μόνο εμείς οι μόνοι παίκτες στην περιοχή, υπάρχουν και άλλοι, οπότε θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Και περιμένουμε πώς και πώς την συνάντηση του Λονδίνου, όπου ο πρόεδρος Καρζάη θα έρθει και θα προσφέρει το πρόγραμμά του. Για να βοηθήσουμε γέμιση ακόμα περισσότερα με τα ε, εξορισμού μακρόπνοη είναι η προσπαθειά μας, βιώσιμη. Και επομένω θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που θα στείλουμε στην περιοχή. Να είμαστε ρεαλιστές. Χρειαζόμαστε χρόνο. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πολλή δουλειά και γι' αυτό η εμπλοκή μας θα είναι μακροπρόθεσμη. Θα πρέπει να είναι και ορατή και έτσι να βοηθήσουμε και ανήλικους και γυναίκες στην περιοχή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Προεδρία για τα ναρκωτικά προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνεκτική απόκριση, δηλαδή ανάπτυξη της υπαίθρου, κράτος δικαίου, κοινωνικό, οικονομικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Είναι όντως πολύ σημαντικά τα μη στρατιωτικά ζητήματα. Έχουμε επιτύχει πρόοδο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το 2002 Ε, καταφέραμε να βοηθήσουμε το 7% του πληθυσμού για υγειονομική περίθαλψη. Τώρα έχουμε φτάσει στο 85%. Αυτό αποδεικνύει το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε. Συμφωνώ με την κυρία που είπε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Οι πόροι είναι αντικείμενο διαχείρισης από τον ΟΗΕ και την Παγκοσμία Τράπεζα και η κατάσταση είναι πολύ καλή. Τον Ιούλιο του 2009 έχω μια έκθεση για τον Ιούλιο του 2009 που καταδεικνύει πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα, ε, πώς ξοδεύονται και τι, ε, ποια είναι η στόχη μας. Συμφωνώ όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και μία από τις προκλήσεις ε, που θα αντιμετωπίσω είναι αυτή. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να ε, σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με τη UPOL. Ε, είχα μια συνάντηση με τον γραμματέα του ΝΑΤΟ, με τον ε, στρατηγό Μακρίσταλ, με τον κύριο Χόλμπρουκ. Μιλήσαμε για το Αφγανιστάν, οπότε ήδη ετοιμάζουμε τη διάσκεψη του Λονδίνου. Και ε, βεβαίω αυτά τα οποία αναφέρθησαν για την περιφερειακή πτυχή του προβλήματο είναι εξαιρετικά σημαντικά. Θέλουμε αυτό το, με το σχεδίο δράση να οδηγήσει σε περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των γειτονικών ε, χωρών εμπορική συνεργασία και πολλά άλλα θέματα. Ε, συμφωνώ λοιπόν απολύτω από αυτό. Η διάσκεψη του Λονδίνου είναι η επόμενη σημαντική καμπή. 28 ε, Ιανουαρίου στο Λονδίνο. Θέματα ασφαλείας, ε, διακυβέρνησης, κοινωνικο-οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Πολύ σημαντικά. Τέλος, Πρόεδρε, είναι θέματα αυτά που εντόπισα και που ανέφερα. Όλα αυτά μπορώ να πω ότι είναι θέματα για τα οποία έχω μακρά πείρα. Thank Έληξε η συζήτηση. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής για τη Λευκορωσία. Πρώτα λαμβάνει το λόγο η κυρία Μάλστρομ του Συμβουλίου.